και δημιούργησε μια πολυφιλετική δημοκρατία στη Νότια Αφρική. Τον χαιρετίζουμε λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφοι. Να ψηφίσουμε τώρα. Πρώτο θέμα λοιπόν είναι η ψηφοφορία για την έκθεση ε, ε, Αλμπερτίνη σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας. Ψηφίζουμε λοιπόν. Έχουμε έτοιμα για ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Σαφές το αποτέλεσμα. 578 ψήφοι υπέρ, 22 ψήφοι κατά, 9 αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Αλβερτίνη. Επόμενο θέμα. Απλουστευμένη διαδικασία λοιπόν, έκθεση μαστάλκα, ανάκτηση διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενικής διατροφής σε αλλοδαπό κράτος. Ψηφίζουμε λοιπόν και σε περίπτωση θα έχουμε ψηφοφορία δοκιμαστικής κλίσεως, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε και αυτό το, αυτή η έκθεση με σαφή πλειοψηφία. 591 ψήφοι υπέρ, 10 κατά, 11 αποχές. Επόμενο θέμα είναι, είναι ψηφοφορία από τις εκθέσεις της κυρίας Γκιόνες, κοινωτικό πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική ελληνική. Πριν ε, ψηφίσουμε θα δώσω το λόγο στην κυρία Γκιόνες, την εισηγήτρια. Πρόεδρε, ήθελα να κάνω δύο σύντομες αναφορές. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης εισηγητές για την συνεργασία τους. Ευχαριστώ και την Κοινοβουλευτική μου Επιτροπή. Ευχαριστώ και